αλλά και την προστασία της κοινωνικής οικονομικής συνοχής των αλλιέων και των οικονομιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλάνα. Θέλω να σας ε, ενημερώσω ότι και η γραπτή δήλωση υπαριθμών 52 σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Down συγκέντρωσε τις υπογραφές μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών από την απλή πλειοψηφία του σώματος και κατόπιν αυτού θα διαβιβαστεί σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση. Ε, ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κούτας, εκ των συντακτών της γραπτής δήλωσης, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω την κυρία Ντανσίλε, την κυρία Νικολάη, τον κύριο Ταραβέλα και την, τον κύριο Ούλμαν για την βοήθεια που έχουν δώσει στην σύνταξη αυτή της έκθεσης και φυσικά και τους συνεργάτες τους, όλους αυτούς που έχουν αγωνιστεί για να καρποφορήσει αυτή η πρωτοβουλία και φυσικά είναι εμβληματική αυτή η πρωτοβουλία το Κοινοβούλιο με τον τρόπο αυτό δείχνει την αλληλεγγύη του με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Down και κάνει ό,τι του αρμόζει για να μπορέσει να διατηρήσει την πολυμορφία στην Ένωση. Τώρα στην ε, ψηφοφορία. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την ε, απλοποιημένη διαδικασία της έκθεσης του κυρίου Σάμπανοτς σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.